Ε, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ελπίζω όλοι να περάσατε ωραίο καλοκαίρι. Ε, από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι από εσά ε, περάσατε καλά και ε, μαυρίσατε και στον ήλιο. Βλέπω ότι ειδικά στο Λουξεμβούργο πρέπει να έχει πολύ ήλιο. Ε, έχετε μαυρίσει περισσότερο από όλου. Α περάσουμε στο σημείο 2 που είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 16 έχει αναβληθεί για μεταγενέστερη συνεδρίαση κατόπιν ετήματος του, της κυρίας Αλβιόλ. Μπορούμε να ε, υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη με την τροποποίηση αυτή και να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης η και 22 Ιουνίου όπως έχουν διανεμηθεί. Ωραία, εγκρίνονται. Επίσης θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω και να καλωσορίσω ε, την κυρία Αντρέα Κρατσιούν στην γραμματεία. Πού βρίσκεστε? Παρακαλώ, σηκωθείτε να σας δούμε. Καλώς ήρθατε. Είσαστε Ρουμάνα νομικός. Χαιρόμαστε που έχουμε νομική ε, εδώ μεταξύ μας. Έχετε και πείρα από ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις στον τομέα της μετανάστευσης, της ενέργειας ε, και του αθλητισμού. Επίσης θα είναι χρήσιμο που η γραμματεία θα έχει μεταφράστρια. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Ε, παρακαλώ συνάδελφοι να είσαστε καλοί μαζί της. Δεν έχουμε κανένα θέμα στα διάφορα και μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία πάνω στην γνωμοδότηση για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πρόκειται για αναδιατύπωση. Ελπίζω να έχετε τοποθετήσει τις κάρτες σας στις συσκευές. Μαρκρέτε, έχεις όμως την κάρτα σου. Όχι. Την έχω, αλλά όχι εδώ, λέει η Okay, we will take your indications. We will take, take... Ωραία, θα, θα έχουμε το νου μας, θα βλέπουμε πώς ψηφίζεις. Ωραία, εξαιρετικά. Ο Ομπάμα πώς το είπε, ε, ε, fueled up and ready to go. Ε, τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 6, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 56, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 58, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Όχι, καταπίπτει 22. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Το δεύτερο τμήμα μόνο ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εβδομήντα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εβδομήντα υπέρ, κατά, αποχές, όχι, λάθος. 77. Η 76 καταπίπτει. Πρέπει να ψηφίσουμε την 75, λέει η πρόεδρος, την 76 μάλλον εννοεί. 76 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Ε, δεν τα χέρια σας. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να την ελέγξουμε. Έναρξη της ψηφοφορίας για την 87, ηλεκτρονική επαλήθευση.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 Από... Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έτσι, για να μας παίρνει ο ύπνος. Λήξη της ψηφοφορίας. Ορίστε, εγκρίνεται κατά μία ψήφο. Το σημειώνουμε. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη της ψηφοφορίας. Για την τροπολογία 98. Λήξη της ψηφοφορίας. Όχι. Λήξη της ψηφοφορίας τώρα. 11 υπέρ, 11 κατά, το οποίο σημαίνει Μαρκρέτε, εσύ πώς ψηφίζεις, υπέρ υποθέτω. Ε, με τη δική σου ψήφο εγκρίθηκε 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας να βλέπω. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 113 έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη της ψηφοφορίας για την 32. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34. όχι, τροπολογία 2. Τροπολογία 2. Διστάμενε από στη γραμματεία. Τροπολογία 2 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 6. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κατόπιν έχουμε προφορική τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 καταπίπτει. Συμβιβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Άλλη μια φορά. 52. Έναρξη της ψηφοφορίας, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Α, να, και η Μαργκρέτε τι ψηφίζει. Απορρίπτεται με την ψήφο της Μάρκαρετ. Τροπολογία 17 και 53 είναι όμοιες ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 18 υπέρ, κατά. Α, και αυτό είναι ασαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση έναρξης ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Όχι καταπίπτει. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και προχωράμε στον επόμενο κατάλογο ψηφοφορίας. Σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, για τις Αναπηρίες. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 18. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, όχι. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Όχι, πρέπει να το ψηφίσουμε, πρέπει. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 23 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ,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 εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να τρέξω στη διάσκεψη των πρόεδρων. Ο Πάλ θα προεδρεύσει τη Τρίτη ψήφου, θα τα πούμε αργότερα. Να είστε καλοί μαζί του παρακαλώ. So if you να συνεχίσουμε λοιπόν. Σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά λοιπόν με την αναφιόρηση του κανονισμού ...211 του 2011. Λοιπόν, συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, να ελέγξουμε. Την τροπολογία 1 ελέγχουμε. Open Close. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όπως λέει η κυρία Όκεν, δεν άλλαξε το πρόβλημα, παρότι άλλαξε ο πρόεδρος, ε, εγώ ψήφισα υπέρ. Γιατί δεν έχει ληφθεί υπόψη. Μάλιστα, εγκρίνεται. Να συνεχίσουμε παρακαλώ τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5. Υπέρ, κατά, σαφές νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Όχι. Καταπίπτει. Ε, 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε ή θεωρείτε ότι εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Εννέα. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, α, κατά πίπτη, ναι, ευχαριστώ. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία... Συμβαστική 3. Α, όχι, όχι. 27. Τροπολογία 27. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καταπίπτει μάλιστα. Πού πάμε? Στην 49, ψήφι υπέρ. 49. αυτό το τμήμα που έχει εδώ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ. Ωχ, καταπίπτει και αυτή. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ούτε 56 πρέπει να ψηφιστεί. Πού πηγαίνουμε. Στην 70. Πού πηγαίνουμε. Συμβιβαστική 7. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 70. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 72. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 74. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εσείς έχετε, ωραία, ψηφίζετε αποχή, εντάξει. Εγκρίνεται το σχέδιο νομοδότη. Πλήρης αυτοσχεδιασμός, σε συγχωρέστε με. Αλλά τουλάχιστον ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, να συνεχίσουμε. Καλό θα ήταν. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να περάσω στη μητρική μου γλώσσα, στα ουγγρικά. Ο 9-es és a 10-es pontokat fogjuk együtt tárgyalni. Είναι το σημείο υπαριθμών 9 και μαζί το σημείο υπαριθμών 10, το οποίο τώρα θα συζητηθούν γιατί ε, αφορούν το ίδιο θέμα οι αναφορές. Καλώς όρισαν οι αναφέροντες. Θα λάβουν τρεις εξ αυτών τον, τον λόγο. Πρώτος ο κ. Ανδρέας Λούζ. Έχετε το λόγο. Τέσσερα λεπτά. Κυρίε και κύριοι, ε, αξιότιμοι βουλευτέ της Επιτροπή αυτής. Το εμπόριο αποτελεί σίγουρα βάση όλων των κοινωνιών. Αλλά πρέπει το εμπόριο να πραγματοποιείται με ίσους όρους και να μην γίνεται εις βάρος κάποιων εμπορικών εταίρων. Η TTIP και η ΣΕΤΑ είναι εμπορικές συμφωνίες ε, όπου με τη βοήθεια ε, προσφυγών ε, των επενδυτών ή με νομοθετική συνεργασία μπορούν να εκβιαστούν τα κράτη και να καταστραφούν οικονομικά. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε με κάθε τίμημα διότι εκατομμύρια ανθρώπων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορέσουν να ζήσουν με τα αποτελέσματα ε, αυτών των ε, συμφωνιών. Το ότι οι διαπραγματεύσεις ε, έγιναν και κλεισμένων των θυρών μας κάνει να αμφισβητούμε την νομιμότητα αυτών των συμφωνιών. Και οι δύο διαδικασίες δεν είναι συμβατές με το γερμανικό σύνταγμα και υπονομεύουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ότι επιτρέπεται η συμμετοχή ε, των λόμπι στην νομοθεσία νωρί και επίση η νομοθετική συνεργασία, αυτό αποτελεί ε, άμεση επίθεση στην κυριαρχία και την δημοκρατία των ε, κρατών αυτών. Ήδη σήμερα υπάρχουν στις Ηνωμένε Πολιτείες γραφεία δικηγορικά, τα οποία ειδικεύονται στις προσφυγές επενδυτών ε, και πετυχαίνουν ε, τεράστια κέρδη για τους πελάτες τους. Υπάρχουν ε, πολλά παραδείγματα για το πού θα μας οδηγήσει αυτή η νομοθεσία δύο τάξεων. Για παράδειγμα, η επιχείρηση Oceana Gold ε, ζήτησε από το Ελσαλβαντόρ 300 εκατομμύρια δολάρια επειδή ε, σταμάτησε ε, κάποια σχέδια εξόριξης. Ή ένα παράδειγμα από τη Γερμανία όπου η Σουηδική Βάτενφαλ ζήτησε 500 δισεκατομμύρια ευρώ επειδή η Γερμανία ήθελε να σταματήσει την ατομική παραγωγή ενέργειας μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα. Θα έχουμε λοιπόν σημαντικές επιπτώσεις. Ε, τα πρότυπα των τροφίμων ε, θα ε, επηρεαστούν αρνητικά. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να σας αναφέρω όλα τα παραδείγματα και όλους τους τομείς που θα επηρεαστούν, αλλά είναι υπερβολικά πολλοί οι τομείς που θα επηρεαστούν. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποσταθεροποιηθεί εάν εφαρμόσει τις συμφωνίες υπό την παρούσα τους μορφή. Το αποτέλεσμα θα είναι απώλεια δημοκρατίας, δημοκρατικό έλλειμμα και βλέπουμε ήδη μία κίνηση προς ε, την ε, άκρα δεξιά στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να παραθέσω τα λόγια του Προέδρου της Ευρωπαϊκής, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πρέπει να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να ενισχύσουμε την δημοκρατική νομιμοποίηση της κοινοτική μεθόδου. Ούτε ο κύριος Ιούνκερ είναι διατεθειμένος ε, να ε, θυσιάσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας, ε, στον κοινωνικό τομέα, στην προστασία των δεδομένων και της πολιτιστικής ποικιλομορφία στον βωμό των ελευθέρων συναλλαγών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και την Τολόρες Ντοράνο Βιθέντε που εκπροσωπεί δύο αναφέροντες που αντίστοιχε αναφορές. Είστε εδώ, μάλιστα. Όταν μια δημοκρατική χώρα όπως η Ισπανία ε, ξεκινά και ολοκληρώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια διαπραγματεύση όσον αφορά μια συνθήκη ελευθερών εμπορίου που είναι τόσο σημαντική όπως το TDIP, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και οπότε γι' αυτό και ζητάμε όσον αφορά το περιεχόμενο σε αυτές τις συνθήκες που αποτελούν το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων ως Ισπανοί δεν μπορούμε να μην, μην διεκδικήσουμε αυτό το δικαίωμα στην πρόσβαση σε αυτές τις συνθήκες και στο περιεχόμενό τους. Έχουν γίνει κάποιες ε, μελέτες όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις και για την TTIP και για την ΘΕΤΑ. Όμως από πλευράς ε, περιβάλλοντος δεν έχουν γίνει μελέτες, οπότε δεν θα μπορούσατε να μας, ε, να μας τα εξηγήσετε γιατί συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιες εκθέσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτών στην Γεωργία. στην Ευρώπη δικαιούμεθα να γνωρίζουμε και να μπορέσουμε να επιλέξουμε αυτό το οποίο τρώμε. Και η εξίσωση της νομοθεσίας μας με την Αμερικάνικη για τη διατροφική ασφάλεια είναι με ένα πισωγύρισμα χωρίς προηγούμενο για τα δικαιώματά μας. Οπότε η Επιτροπή και η Επιτροπή δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν εκθέσεις για το ποιε είναι οι συνέπειε των συνθήκων για του εργαζόμενου και για τη δημοσία υγεία από την άλλη μεριά. Εάν το ISDS ε, ισχύσει τότε μπορούν να ζητήσουν οι πολυεθνικές να αλλάξει το κράτος την νομοθεσία. Αυτά όσον αφορά τι ισχύει μετά την TTIP. Επομένω, τώρα εδώ πέρα έχουμε ένα κείμενο για το περιβάλλον και τη σχετική νομοθεσία. Έχουμε επίση το Ecologic Institute που έχει επισημάνει του κινδύνου εδώ στι Βρυξέλλε και ζητεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εφαρμόσει αυτό το σύστημα επίλυση διαφορών. Επομένω, δεν έχουμε διαφάνεια. Προχωρούμε αντίθετα από τις ε, μελέτες αυτές που αξιολογούν τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν για τον κόσμο οι κατάλληλες πληροφορίες. Όμως το site της web όσον αφορά για το TTIP αλλά και όσον αφορά την ΦΕΤΑ, ΣΕΤΑ δηλαδή τη Συμφωνία για Εμπόριο και Υπηρεσίες θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε το σύνολο του κειμένου, να μπορούμε να τα μελετήσουμε και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις ε, συνέπειες. Έτσι υπάρχουν εγγυήσεις για τη συμμετοχή του πολίτη και εγγυήσεις διαφάνειας. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Δεν γνωρίζω το όνομα του τρίτου. Αναφέροντας μόνο τα αρχικά έχουμε. Παρίσταται. RZ. Ροζίτα είναι τα αρχικά σας. Λίγα και μόνο μας έχετε δώσει τόσο ώστε να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Οπότε θα σας παρουσιάσω απλώς μια μικρή περίληψη από όλα αυτά τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτο ζήτημα Σήμερα η Αφρικανική Ήπειρος έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. Μόνο το 5%, το 5% λέω, αυτού του πληθυσμού μεταναστεύει. Πρώτα, για 65 εκατομμύρια. Αυτοί κατευθύνονται προς την ε, Ευρώπη και συγκεκριμένα προς την Ιταλία. Πρώτο μας έτοιμα ε, Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν τις συνθήκες του Μαστρίτ, δηλαδή ε, εδώ και 25 χρόνια τελικά καθόρισε με ακρίβεια κάποιους κανόνες όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα για τα 27 κράτη-μέλη. Επίσης δεσπίστηκαν συγκεκριμένες κυρώσεις κατά όσων διαβαίνουν τα σύνορα χωρίς άδεια. Πρόκειται για μια αρχή που ισχύει χωρίς καμία αμφισβήτηση όσον αφορά τα σύνορά μας. Δεύτερο ζήτημα. Τα σκάφη όλων των χωρών μελών μεταφέρουν όλους αυτούς τους ε, μετανάστες αυτούς που τους περισυλλέγουν από τη θάλασσα. Η Ιταλία μόνη της δεν μπορεί να το κάνει αυτό και να υποστεί το σχετικό κόστος. Τρίτο αίτημα. Οι διακινητές και όσοι είναι ύποπτοι για τέτοιες ε, ενέργειες να φυλακίζονται και έτσι να αποτρέπονται οι επόμενοι. Αυτοί όλοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το σκάφο του προς τούτο και να καταστρέφονται τα σκάφη αυτών των διακινητών έτερων. Χρειάζεται έλεγχος συνεχής όσον αφορά τι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουν κατηγορηθεί από την Frontex ότι συμπράττουν με τους διακινητές. Επίσης, με δεδομένο ότι οι, οι βουλευτές θα πρέπει να φροντίζουν τα δέοντα. Θα πρέπει να φροντίζουν για την ευημερία των Ευρωπαίων. Θα πρέπει να κάνουν κάτι για αυτά τα αιτήματά μας θα πρέπει επίσης να ματαιωθούν να αναφιωθούν αυτές οι διατάξεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα κάποιων προϊόντων μας. Έχουμε καταλήξει να έχουμε κρασί που δεν είναι από σταφύλια και σοκολάτα η οποία δεν προέρχεται από το κακά. Έχουμε τυρί το οποίο μπορεί να παραχθεί χωρίς να έχει μέσα τυρίνη καζέινη. Ε, και από γάλα σκόνια. Όλα αυτά θέτουν κινδύνο την υγεία των καταναλωτών. Και μόνη των ιδίων που με ακούτε. Έκτο αίτημα. Σε σχέση με τη συμφωνία TTIP και το ΣΕΤΑ, χρειάζεται να ανακληθούν και η συμφωνία με τον Καναδά. Και όπως έχει, πει ο πρόεδρος μας ε, Ρομπέρτο Κάλβο ότι όλα αυτά είναι ένα δωράκι προς τις πολυεθνικές της βιομηχανίες των ειδών διατροφής. Και όλα αυτά είναι μεγάλη ζημιά για την Ιταλία επίσης. Δεν θα πρέπει να διευκολύνεται η Κίνα αλλά και άλλες αντισώμενες χώρες γιατί αυτό αφορά κάποια δικαιώματα συνδικαλιστικά. Είναι απαράδεκτο να προβαίνουμε σε συμφωνίες εμπορικές στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης με κάποιες τέτοιες χώρες όπου υπάρχουν εργαζόμενοι παιδιά που είναι και οκτώ χρόνων. Όλα αυτά είναι καταστροφικά για την ε, υγεία του, αλλά επίσης και για το συνταξιοδοτικό. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και τους τρεις αναφέροντες. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρενίτα Μπάσκαρ, παρακαλώ, για το TTIP και τη ΣΕΤΑ. Ευχαριστώ. μου ζητήθηκε να σας μιλήσω για το πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συμφωνία TTIP και ΣΥΤΑ. Θα κάνω αυτό το σύντομο απολύσμα και μετά θα δώσω απαντήσεις σε ορισμένα από τα στήματα τα οποία έθεσαν οι αναφέροντες. Αυτό που θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή είναι ότι οι διαπραγματεύσει ε, για την συμφωνία TTIP ε, έχουν ανασταλεί από τότε που άλλαξε η κυβέρνηση στι ΗΠΑ. Οι προτεραιότητες και τα συμφέροντα της ε, νέας κυβέρνησης ε, για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ασαφέστατα και τα μηνύματα τα οποία έχουν δοθεί είτε δημοσία είτε ε, με άλλους τρόπους είναι ότι η κυβέρνηση ασχολείται με άλλες ε, διαπραγματεύσεις τη Συμφωνία Ναύτα εξετάζει και εξετάζει και ζητήματα που έχουν ανακύψει με άλλους διμερείς εταίρους όπως είναι η Κίνα οικονομικό σκεπτικό για την έρξη των διαπραγματεύσεων μπορεί να μην είναι θετικά τα μηνύματα αλλά το ε, σκεπτικό ισχύει πρόκειται για τη συμφωνία μεταξύ δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους άρα από οικονομικής πλευράς έχει νόημα να γίνει προσπάθεια εξομάλυνσης των εμποδίων να γίνει προσπάθεια ε, να υπάρξει μια ισορροπημένη και αμοιβαίως εποφελή συμφωνία. Και βέβαια δίνεται ευκαιρία και για εμάς από κοινού να χαράξουμε, να διαμορφώσουμε τους παγκόσμιους κανόνες. Ό,τι αφορά τώρα την ίδια την διαπραγμάτευση, πριν διακοπή, πριν ανασταλεί, υπήρχε πρόοδος σε πολλούς τομείς, αλλά υπήρχαν και σημαντικές διαφωνίες με τις ΗΠΑ αποκλήσει απόψεων σε τομεί όπως είναι οι δημόσιε προμήθειε, πολύ σημαντικό τομέα οικονομικού ενδιαφέροντο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν προβλήματα και στον τομέα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είχαμε βαθιές διαφορέ, δεν γεφυρώθηκε το χάσμα. Τα μηνύματα που στέλνει η νέα κυβέρνηση βέβαια πηγαίνουν ακόμα πιο πολύ προ την αντίθετη κατεύθυνση. Άρα οι πιθανότητε επανέραξη των διαπραγματεύσεων τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον είναι πάρα πολύ ε, ε και η Επιτρόπος Μάλστρομ ξεκαθάρισε τη θέση της ε, και είπε ότι θα πρέπει πριν ξαναξεκινήσουν οι παρτέρες να γίνει μια πολύ ε, αναλυτική συζήτηση με την Αμερικανική πλευρά για να έχουμε λάβει διασφαλίσεις ότι μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος ε, σε αυτές τις πραγματές ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά για μια ισορροπημένη συμφωνία. Θα ήθελα να αναφέρω τώρα, αν μου επιτρέπετε, κάποια σχόλια που αφορούν τα ζητήματα που έθεσαν οι αναφέροντες. Ένα ζήτημα ήταν το ζήτημα της διαφάνειας. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι πράγματι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP κατά κάποιο τρόπο ε, σημαδεύτηκαν από μια τομή ε, σε ό,τι αφορά το πώς ε, χειριζόμαστε τα έγγραφα. Επειδή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τελικά ε, προβήκαμε σε μία εκβάθρον μεταρρύθμιση του συστήματος και του τρόπου τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή με την κοινή γνώμη, δημοσιοποιούμε τις θέσεις μας, τα κείμενα τα οποία έχουμε διαπραγματευτεί. Για να έχουμε λοιπόν επαφές με την κοινότητα των πολιτών, έχουμε και μία ομάδα συμβουλευτική η οποία συναντάται και γίνεται και τακτή ενημέρωση. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε γιατί αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί διαπραγματεύσει. Τώρα, παρομοίω το γεγονό ότι όλε οι θέσει και όλα τα κύματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιοποιήθηκαν, δημοσιεύθηκαν, δεν νομίζω ότι φαίνεται από τίποτε ότι δεν ε, τηρούμε τις, ε, τα πρότυπα για τα οποία, ε, από στα οποία αποδίδουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είτε για τα τρόφιμα, ότι έχει παραβιαστεί κάποια γραμμή. Ήδη πρέπει να σας πω ότι πριν ξεκινήσει να ισχύει οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να δώσει τη συμφωνία μου, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι πάντοτε πρέπει να γίνεται. Επίσης ακούστηκαν πολλά σχόλια για το ISDS. Το ε, σύστημα επίλυσης ε, των ε, διαφορών στο πλαίσιο του Τύπη και ξεκίνησε μια τεράστια μεταρρύθμιση λόγω των διαπραγματεύσεων. Περάσαμε σε ένα σύστημα το οποίο είναι πιο σαφές, πιο διαφανές. Υπάρχει πλέον ένα μόνιμο δικαστήριο, έχει συγκροτηθεί για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων που υπήρχε, είχε δημιουργήσει μάστιγα στα παραδοσιακά νομικά συστήματα. Και σε ό,τι αφορά την ηθική της διαδικασίας έχουμε ενισχύσει αυτές τις πτυχές. Έγινε και μια πολύ μεγάλη μελέτη, είναι η μελέτη αντικτύπου βιωσιμότητας, έχει δημοσιοποιηθεί νωρίτερα φέτος για το TTIP και παρότι έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις θα βρείτε ένα σημαντικό τμήμα στην ε, έκθεση αυτή που αφορά ε, το περιβάλλον ε, και το, την υγεία, τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ΣΕΤΑ, προσωρινά Ισχύει η Συμφωνία 21 ε, Σεπτεμβρίου ε, τίθεται προσωρινά σε ισχύ μετά την υπογραφή της ΕΤΑ ε, στην διάσκεψη κορυφής τον Οκτώβριο του 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά και επίσης έδωσε και σύμφωνη γνώμη το Κοινοβούλιο για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Η ΣΕΤΑ είναι αναγνωρισμένα μία από τις πιο σύγχρονες συμφωνίες. Ο Κάναδας ε, είναι ένας από τους πιο στρατηγικούς μας εταίρους, ιδίως σε ασταθείς καιρούς. Αυτά έχω να πω και αν υπάρχουν ερωτήσεις μπορώ να επανέλθω. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τώρα το έγγραφο για την ΤΙΣΑ, να δώσω το λόγο στον κύριο Κίνερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αναφέροντες ε, για το ενδιαφέρον τους ε, και για τις απόψεις που εξέφρασαν. Πολύ σύντομα για την ΤΙΣΑ. Ισχύει ακριβώς ότι εξήγησε η Ειρήνητα για την TTIP. Οι διαπραγματεύσεις ε, βρίσκονταν σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωσή τους σε τέλη ε, του προηγούμενου έτους όταν ε, πραγματοποιήθηκαν οι προεδρικές εκλογές ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό οδήγησε σε πάυση των διαπραγματεύσεων για την ΤΙΖΑ. Δεν έχει υπάρξει έκτοτε καμία δραστηριότητα. Ούτε έχουμε λάβει κανένα μήνυμα από τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα ήθελαν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις σύντομα. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά, οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, είναι ε, προ συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι, θα, διότι είμαστε πολύ ισχυροί στον τομέα των υπηρεσιών και πολύ σύντομα να, επανα, να, να απαντήσω στα όσα άκουσα για τις υπηρεσίες. Καταρχάς, η εντολή μας είναι δημοσίως διαθέσιμη όλες οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα έγγραφα που έχουμε λάβει από τους άλλους εταίρους, τα οποία δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε, έχουν διαβιβαστεί στα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου έχουν συζητηθεί στο σωστό πλαίσιο. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάρος Λαβαλέσα, εκ των μελών πρώτος. Συγγνώμη που θα τα πω έξω από τα δόντια, αλλά νομίζω ότι το να συζητούμε αυτές τις αναφορές στην παρασχρονική στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Καταλαβαίνω ότι οι αναφορές αυτές αναφέρονται σε πολύ σημαντικά ζητήματα TTIP, ε, SETA, ΤΙΣΑ. Πολύ σημαντικές ε, συμφωνίες για όλους μας. Όμως, Αν κάνουμε μια θεματική υποδιέρεση αυτών των συμφωνιών, ε, των αναφορών, βλέπουμε ότι η ΣΕΤΑ ε, τέλειωσε, ψηφίστηκε. Κάνα δύο μήνες πριν δώσαμε σύμφωνη γνώμη. Και το αποχείρημα που άκουσα από τους αναφέροντες ήταν η μη πρόσβαση στα έγγραφα, κάτι το οποίο δεν αληθεύει, γιατί ψηφίστηκε και είναι διαθέσιμο το έγγραφο. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο. Τώρα, σε ό,τι αφορά, επομένως, σε ό,τι αφορά τη ΣΕΤΑ, νομίζω ότι τι ε, σχετικές αμφώσεις πρέπει να τι κλείσουμε αφού η συμφωνία έχει ψηφιστεί. Τώρα, για τι άλλε δύο τα πράγματα είναι διαφορετικά, TTIP και ΤΙΣΑ. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτέ τι συμφωνίε, αλλά πριν τη διαδικασία επικύρωση όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει. Αλλά και η TTIP και η TISA έχουν ανασταλεί προ το παρόν. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο. Δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο διαθέσιμο. Και ένα κανόνα των διαπραγματεύσεων ήταν και είναι πάντοτε Nothing is agreed until everything is agreed. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο αν δεν έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Άρα δεν μπορούμε αν δεν έχουμε ένα έγγραφο στο οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε, να συζητήσουμε. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στι αναφορέ αυτέ μόνο όταν θα έχουμε ένα έγγραφο ενώπιον μα και να συζητήσουμε τα πολύ σημαντικά ζητήματα που θέτουν. Για την ΤΙΣΑ και την ΤΙΤΙΠ λοιπόν αυτό το οποίο προτείνω είναι να μπουν στον κατάλογο των θεμάτων Β. Ευχαριστώ κύριε Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες γιατί έθεσαν αυτά τα σημαντικά θέματα τα οποία δεν απασχολούν μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απασχολούν εδώ και πολλά χρόνια όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Δεύτερον, η TTIP, η ΣΕΤΑ, και η TISA έχουν ένα μοντέλο συγκεκριμένο. Και μπορεί ναι μεν η TTIP και η TISA να έχουν ανασταλεί, αλλά η αντίληψη και οι λογικές μέσα από το μοντέλο που έχει διαμορφωθεί συνεχίζουν να υπάρχουν και σε άλλες διαπραγματεύσεις. Επομένως έχει αξία να συζητήσουμε. Και να συζητήσουμε τι. Πρώτον, ότι μέσα από το διεθνές εμπόριο ουσιαστικά δημιουργείται ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα γιατί επί, τους, επί της ουσίας οι λαοί και τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να παίξουν σοβαρό ρόλο. Δεύτερον, υπάρχει ένα έλλειμμα δικαστικής προστασίας, διότι όλα αυτά τα μοντέλα, τα καινούργια των συμφωνιών αυτών, δημιουργούν ε, δικαστήρια ειδικά, δικαστήρια διαιτησία στην πράξη και ακυρώνουν τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των κρατών μελών. Τρίτον, όλες αυτέ οι συμφωνίες δίνουν εξουσίες σημαντικές, κυρίω στι πολιεθνικές οι οποίε μπορούν ε, να ασκήσουν αγωγέ αποζημίωση κατά των κρατών μελών. Τέταρτον, επί της ουσίας διαλύουν την οικονομία και στηρίζουν κυρίως τις μεγάλες πολυεθνικές, είτε είναι αμερικανικές, είτε είναι ευρωπαϊκές, είτε είναι κινέζικες, αλλά διαλύουν τις τοπικές οικονομίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον διαλύεται τελείως η γεωργία και αυτό κάτι το έχουμε δει επί του πρακτέου. Καμία προστασία στη δημόσια υγεία και στους καταναλωτές. Διάλυση και απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Και εξαφάνιση αυτού που ονομάζουμε προϊόντα ονομασίας προέλευσης, POP, όπως είναι η φέτα, η οποία πλέον δεν έχει καμία προστασία λόγω της κύρωσης της ΣΕΤΑ. Άρα λοιπόν τα θέματα έχουν αξία, είναι σημαντικά. Και να απευθυνθώ λοιπόν προς την Επιτροπή και να πω το εξή, Έχει εκδοθεί πριν λίγο καιρό μια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Σιγκαπούρης. Και τι έχει πει. Ότι η συμφωνία αυτή είναι μεικτή Δηλαδή ότι υπάρχουν συμφωνίες όπου υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να αποφασίσει, αλλά όταν είναι μικτής φύσεως οι συμφωνίες, για να ισχύσουν χρειάζεται και η κύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια. Ποιο είναι όμως το τρίκ το οποίο έγινε με τη ΣΕΤΑ. Η ΣΕΤΑ έχει τεθεί, όπως είπε και η Κομισιόν, παράνομα κατά την άποψή μας και αυτά δεν τα λέω μόνο εδώ, τα έχω πει επανειλημμένα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παράνομα έχει τεθεί σε εφαρμογή προσωρινή από τις 21 Σεπτεμβρίου. Γιατί? διότι για να ισχύσει μία συμφωνία μεικτή, όπως είναι η περίπτωση της ΣΕΤΑ, πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Επομένως δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή παρά μόνο όταν κυρωθεί από τα 28 κράτη. Τι αποφάσισε όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρανόμως και η Κομισιόν και η πλειοψηφία των κρατών ότι θα τεθεί λέει σε προσωρινή ισχύ και αν κάποιο κοινοβούλιο μετά από τρία-τέσσερα χρόνια δεν το επικυρώσει τότε προφανώς δεν θα ισχύσει η συνθήκη. Αυτό είναι παραβίαση των συμφωνηθέντων, παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, παραβίαση των δικαιωμάτων των ε, εθνικών κοινοβουλίων. Και έτσι λοιπόν είναι όλα τα θέματα στο τραπέζι. Άρα απαντώντας και στον συνάδελφο Βαλέσσα να πω το εξή. Πρώτον, ότι όλες οι αναφορές αυτές πρέπει να, να κρατηθούν ανοιχτές. Για δύο λόγους. Δεν έχει σημασία αν ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο η ΣΕΤΑ και αν έχει παρανόμως προσωρινή εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτό γιατί υπάρχει μια διαδικασία επικύρωσης στα εθνικά κοινοβούλια, άρα είναι ανοιχτός ο δημοκρατικός διάλογος. Επομένως για τη ΣΕΤΑ είναι δεδομένο ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές. Για την TTIP και για την, ε, και για την ε, TISA επίσης πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει τις συμφωνίες. Απλά ο Τραμπ ανέτρεψε τις προσπάθειες που έκανε ο Ομπάμα και η πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή θέλουν, τα κείμενα υπάρχουν και τα κείμενα αυτά είναι σε αυτά στα οποία διαφωνούν και οι αναφέροντες και εμείς. Επομένως κλείνω κύριε Πρόεδρε, όλες οι αναφορές πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές. Δεύτερον, να αποσταλεί ενημερωτικό σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αναφορές των αναφερόντων οι οποίοι διαφωνούν με τη διαδικασία της ΣΕΤΑ και άρα προφανώς είναι υποστηρικτικές προς την μη κύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια. Άρα να ενημερωθούν όλα τα εθνικά κοινοβούλια για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στανόσκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αναφέροντες των αναφορών στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης και ιδιαίτερα τους παρόντες. Βλέπουμε ότι πολλοί τους υποστηρίζουν. Είδαμε και πόσες αναφορές υποβλήθηκαν για το ίδιο θέμα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση η οποία ξεκίνησε το 2013 κατά την συζήτηση των διαπραγματεύσεων αυτών. Πραγματικά τότε δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα των εκλογών στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εμάς μας απασχολεί το θέμα της διαφάνειας, της έλλειψης της διαφάνειας. που αποτελούν και την ουσία των προτάσεων αυτών. Είμαστε κατά λοιπόν, και της ΣΥΤΑ και της TTIP. Ναι, πράγματι βελτιώθηκε η διαδικασία εν μέρη, χάρη στην ανησυχία και τις διαμαρτυρίες του κοινού. Συμφωνώ απολύτως με τα επιχειρήματα του κυρίου Μαριά, γιατί δηλαδή θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές και όσον αφορά την TTIP και την TISA, καθώς και όσον αφορά την ΣΕΤΑ. Ε, να κρατήσουμε ανοιχτές τις αναφορές αυτές και ευχαριστώ και πάλι τους αναφέροντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι λείπει από τη συζήτησή μας μέχρι τώρα. Το πλαίσιο, γιατί ε, επανήλθαν στην Επιτροπή μας αυτές οι αναφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το ανέφερε αυτό. Η απόφαση του ΔΕΚ να σταματήσει η TTIP ε, είναι ε, μεγάλη σημασία σε όσον αφορά το γιατί συζητάμε ακόμα τις συμφωνίες αυτές. Θα ήθελα να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προβλέπει να αντιμετωπίσει την απόφαση του δικαστηρίου να επιτραπούν ECI στις συμφωνίες αυτές, διότι αυτό ε, έχει να κάνει με την αντίδραση του κοινού στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Εάν δεν θέλουμε να καταλήξουμε εκατομμύρια πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συσπηρωθούν και να ε, αμφισβητήσουν την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στους αναφέροντες ε, θα ήθελα ε, να πω κάτι σε συνέχεια των παρατηρήσεων της κυρίας Δανόκα. Έχουν, έχει γίνει πολύ πρόοδος. Ε, ευχαριστώ λοιπόν και εσάς και τους πολλούς ανθρώπους που υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πολλούς που έχουν συζητήσει με ευρωβουλευτές σχετικά με θέματα εμπορικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό οι εμπορικές ε, διαπραγματεύσεις να πραγματοποιούνται με όσο γίνεται πιο ανοιχτό και διαφανή ε, τρόπο. Ε, ε, ήμουν διαπραγματεύτρια συνδικαλιστικών οργανώσεων και πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο και κλεισμένων των θυρών, διότι αλλιώ δεν υπάρχει περιθώριο ευελιξία στις διαπραγματεύσεις, αλλά πολύ μεγάλο μέρος θα πρέπει να πραγματοποιείται δημοσίως. Πολλά λοιπόν ε, έχουν αλλάξει στην πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πόσα ε, έγγραφα πια διατίθενται δημοσίως. Πρόβλημα όμως έχουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου ακόμα και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από το Συμβούλιο να δημοσιεύσει έγγραφα όπως είναι οι διαπραγματευτικές εντολές, ε, τα κράτη-μέλη έχουν μπλοκάρει τη δημοσίευση αυτών των εγγράφων. Νομίζω ότι ως Επιτροπή χρήσιμο είναι να στείλουμε επιστολή στο Συμβούλιο, θυμίζοντα του πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια στι εμπορικέ διαπραγματεύσει, διότι αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο τι προσπάθειε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πετύχουμε περισσότερη διαφάνεια στι συμφωνίε αυτέ, αλλά και τις προσπάθειες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να πιέσει το Συμβούλιο να δημοσιεύσει ε, τα έγγραφα. Για μένα λοιπόν η διαφάνεια είναι το βασικό θέμα εδώ, διότι είναι απολύτω απαραίτητη για την εμπιστοσύνη του κοινού. Ε, να απαντήσω όμως σε κάποιες παρατηρήσεις των αναφερόντων, ιδιαίτερα όσον αφορά το ISDS. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Επίτροπη χρησιμοποιεί ε, ε, ως εναλλακτικές ε, ε τους όρους ISDS και ISDS. Αυτό δηλαδή που παρουσιάστηκε ως τεράστια μεταρρύθμιση του ISDS απλά αποτελεί μια μικρή ρύθμιση. Ε, συνεχίζουμε να έχουμε το πρόβλημα ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ε, έχουν προνομιακή πρόσβαση στη δικαιοσύνη που δεν έχουν οι εγχώριες εταιρείε. Ε, και αυτό όχι μόνο είναι θέμα απλής δικαιοσύνης, όλοι δηλαδή έχουν ίση πρόσβαση και δίκαιη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αλλά θέτει και θέματα συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη πολύ χαρακτηριστικό είναι στην ε, περίπτωση της Σιγκαπούρης που είδαμε στο ΔΕΚ, είναι ότι το δικαστήριο ρητά είπε ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ε, συμβατότητα του ISDS και του ICS με την ε, Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Και αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί προτού συναυθεί οποιαδήποτε συμφωνία που να συμπεριλαμβάνει ISDS ή το νέο σύστημα ICS. Όσον αφορά τα πρότυπα, νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι όσον αφορά τον Καναδά έχουμε καλά νέα. Ως αποτέλεσμα της πίεσης του κοινού και της πίεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα στην στον Καναδά. Ε, ο Καναδάς έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και αυτό αποτελεί αποτέλεσμα εκστρατείας στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε, όλη τη... και σε όλον τον Καναδά για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Νομίζω ότι όσον αφορά την συμφωνία ΣΥΤΑ, αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη και αποτελεί αποτέλεσμα των διαμαρτυριών, των εκστρατιών. Σας ε, καλώ λοιπόν να συνεχίσετε να διαμαρτύρεστε, διότι έτσι πετυχαίνουμε τα βήματα πρόοδου. Να αναγνωρίζουμε όμως και ε, τα θετικά που προκύπτουν, διότι αν δεν έχουμε νίκες είναι εξαντλητικό το να συνεχίζει κανείς να διαμαρτύρεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτές τις μικρές νίκες για να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για πιο δίκαιη και πιο ε, διαφανή εμπορική πολιτική ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προοδεύουμε όμως και προοδεύουμε μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Εύη, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και αυτές οι αναφορές θα πρέπει να μείνουν ανοιχτέ γιατί πρέπει χάρη. Όσον αφορά την μόνο από πλευρά ευρωπαϊκής κύρωσης της ε, ΣΕΤΑ έχουμε το θέμα της κύρωσης από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει εν ώψη αυτού να ενημερωθούν τα Εθνικά Κοινοβούλια όπως είπε ο Μαριάς και για το ΣΕΤΑ τι ενημέρωση έγινε, λευκές σελίδες για κάποια κεφάλαια. Δεν βρήκαμε να έχει κλειστή συμφωνία. Γι' αυτό και είναι λευκές οι σελίδες. Να, για παράδειγμα το κεφάλαιο που αφορά τα φυτοϊγειονομικά και υγειονομικά. Κάτι που έχει παραπενθεί το θέμα στην συγκρισιμότητα των προϊόντων μιας και της άλλης πλευράς. Τι θα γίνει στο μέλλον, ποιο θα τα κρίνει όλα αυτά, κάποιοι τρίτοι, κάποιοι φορεί, κάποιες επιτροπές, κοινέ υπέρ εθνικές. Και είναι αυτός ο οργανισμός ε, ρυθμιστικών, κανονιστικών αρμοδιότητων. Μα ποιος θα τα ε, καταρτήσει όλα αυτά, πού είναι η διαφάνεια, πού είναι η συμμετοχή δημοκρατική των πολιτών. Επομένως, τόσο σημαντική νομοθεσία θα ανατεθεί στα χέρια κάποιου που δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Είναι θέματα επίσης υγεία μας. Προτύπουν ασφάλειας. Όλα αυτά τίθενται να αμφιβόλο. Πολύ απλά είναι τα γνωστά στοιχεία που υπάρχουν, τα οποία με κατέπληξαν όταν τα άκουσα. Έχουμε 93 θανάτους ετησίως από το θέματα διατροφής. 3.000 είναι το αντίστοιχο νούμερο για τη ΣΥΠΑ. Δεν χρειάζεται να σας πω πώς συγκρίνεται ο πληθυσμός ο ένας με τον άλλο. Έτσι καταλαβαίνει κανείς πόσο διαφορετικά είναι τα μοντέλα που κυριαρχούν στη μίξη στην άλλη πλευρά. Ε, το δικό μας είναι πολύ πιο ασφαλές. Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι αυτοί οι κανόνες, αυτά τα πρότυπα που έχουμε κατοχυρώνονται και θα τηρηθούν από τις μεγάλες εταιρείες. Επομένως, να υποστηρίξουμε την προσπάθεια του αναφέροντα από τον ευχαριστούμε που ήρθε. Για τις ΜΜΕ επίσης αυτό είναι μια ευκαιρία. Η ΜΜΕ που είναι το 50% του ιστού μας, του κοινωνικο-οικονομικού, τουλάχιστον έτσι στην Ιταλία, δεν πρόκειται να ωφεληθούν από αυτές τις συμφωνίες. Με κατακλείδω να σας πω ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι να γκρεμίζουμε την εσωτερική αγορά, να γκρεμίζουμε τις ε, ε, ανταλλαγές τις ενδοευρωπαϊκές και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ωφελούμε τις υπερατλαντικές σχέσεις αυτούς δηλαδή που σήμερα έχουν την ισχύ έχουν τις δυνατότητες τις παραγωγικές να έχουν ε, τεράστια παραγωγή και ένα μεγάλο εμπορικό δίκτυο. Απλώς τους αυξάνουμε τα κέρδη. Καταστρέφουμε τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις. Να μείνουν ανοιχτές οι αναφορές. Πρόεδρε, με επιστολή να ενημερωθούν όλα τα κατημέλη για αυτές τις αναφορές. Κυρίως Εν ώψη του ότι του αμέσω επόμενους μήνες τα κράτη-μέλη πρόκειται να προβούν στη διαδικασία κύρωσης σε εθνικό επίπεδο γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ε, ανησυχίες για το θέμα αυτό από τον κόσμο. Είμαι μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και έχω παρακολουθήσει και πολεμήσει κατά των συμφωνιών ΣΥΤΑ και τι τα τελευταία χρόνια και χαίρομαι που βλέπω τόσες πολλές αναφορές. Χαίρομαι που βλέπω και τους αναφέρονται σήμερα εδώ. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα καταπραγητικά κάποια σχόλια της ε, Κομισιόν και του κύριου Κίνερα από τους βασικούς διαπραγματευτές ε, με απογοητεύουν γιατί ε, δεν ε, έχει πεθάνει η TTIP ή απλά πήκε στον πάγο και θα μπορούσε η Κομισιόν να διαπραγματευτεί. Απλά υπάρχουν άλλες διαπραγματεύσεις που την απασχολούν. Ο πρόεδρος Γιούνκερ φαίνεται ότι θα ανακοινώσει σύντομα μία δέσμη πολλών νέων διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα και παραμένουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αδιαφανέστατες, ε, δεν γνωρίζουμε τίποτα και το μόνο που μπορούμε ως Κοινοβούλιο να κάνουμε είναι να πούμε ναι ή όχι. Και η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανωθήκαμε από μόνοι μας ε, και για κάποια πολύ ε, σημαντικά ζητήματα ε, δεν υπάρχουν καν ψηφίσματα τώρα σε ό,τι αφορά το SDS. Δεν άλλαξε κατ' ουσίαν. Ένα μποτοξάκι του κάνανε. Και χαίρομαι πολύ που ζητάει το Βέλγιο ε, την γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμβατότητα του SDS με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη που ίσως τελικά βάσει, βάλει ένα φρένο στη δικασία επικύρωση και μακάρι να γίνει αυτό. πρέπει να πω ότι είχαμε 3,5 εκατομμύρια υπογραφές, αλλά τις αγνόησα όταν συζητούσαν τη συμφωνία ΣΕΤΑ. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό και αλλά όλο και μεγαλώνει. Διευρύνεται το χάζο μεταξύ ε, των ομαθών και των απλών πολιτών και πραγματικά πρέπει να τεθεί ένα τέρμα. Θα ήθελα να ακούσω την Κομισιόνα. Ε, πώς θα το κάνει αυτό και θα, θα, θα ακούσει επιτέλους τους αναφέροντες. Ελπίζω να ακουστούν οι αναφέροντε. Παρακαλώ την Επιτροπή σα να κρατήσει ανοιχτέ τι αναφορέ. Επίση, η δική μου πολιτική ομάδα πάντοτε ζητούσε τη διοργάνωση μια δημόσια ακρόαση για τι συνθήκε τι συμφωνίε, μάλλον τι άλλε και για την παγκόσμια εμπορική πολιτική εν γέννη. Ευχαριστώ. Σένα Ροντρίγκεθ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούστε, και εγώ θέλω να εκφράσω την απόψή μου, η οποία είναι να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες αναφέρσεις που ήρθαν εδώ, παρά την έλλειψη διαφάνειας που υπήρξε σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις και που παραμένει. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το λέω στην Κομισιόν ότι εξακολουθεί να είναι ε, σε φάση διαπραγμάτευση πολλέ φορέ. όπω αυτή με την Χιλή, την Ιαπωνία, ε, το Μαρόκο, τη Νέα Ζηλανδία κτλ. λοιπά Και πολλοί βουλευτέ ε, δεν έχουμε καν πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία είναι υποδιαπραγμάτευση αυτό, για αυτές τις συμφωνίες που είτε είναι σε ισχύ και άλλες που δεν έχω αναφέρει ακόμη. Ξέρουμε όλοι, υπάρχουν πολλές, πολλές συμφωνίες που διαπραγμάτευση και δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε στο Κοινοβούλιο για τους βουλευτές εν γέννη και ούτε και για τους πολίτες όσο μάλλον. Κατά δεύτερον, πραγματικά είναι κοροϊδία να μας λέτε ότι τίθεται προσωρινά σε εφαρμογή η Συμφωνία ΣΕΤΑ χωρίς να έχουν αποφανθεί τα, ευρωπαϊκά κοινοβούλια, τα, συγγνώμη, τα εθνικά κοινοβούλια συνολικά. Συμφωνώ με πολλά από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Αυτό που θέλω όμω να πω είναι, δίνοντας κάποια νέα επιχειρήματα, μας ανησυχεί τα μάλλα κλιματική αλλαγή και φαίνεται τελικά ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε, να εφαρμόσουμε κάποιες εμπορικές συμφωνίες που θα φέρουν ε, κοντά μας πολλά ε, προϊόντα ε, που θα έρχονται κάνοντας τον κύκλο του πλανήτη. Μιλάμε δηλαδή για μεγάλες εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων και μεγάλη μόλυνση. Πού βρίσκεται εδώ η αρχή της προφύλαξης επίσης, αυτό θέλω να ρωτήσω σε όλες αυτές τις πραγματεύσεις και για να ολοκληρώσω θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι πρόκειται για επίθεση κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρέπει να πούμε ότι είναι και μια επίθεση κατά της μικρής κλίμακας ε, ε, γεωργίας, δηλαδή των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών που διαπραγματεύονται. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει με αυτέ τι συμφωνίε. Ζητώ από την Επιτροπή Αναφορών να παραμείνουν ανοιχτέ πράγματι όλε αυτέ οι αναφορέ και ζητώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις διαπραγματεύσεις όλες αυτές να τις αναστείλει και να πάψουν να ισχύουν αυτές οι συμφωνίες που το μόνο που κάνουν είναι να ευνοούν τις μεγάλες πολυεθνικές, το μεγάλο κεφάλαιο. Και οι περισσότεροι από τους συμπολίτε μας, οι λαϊκές τάξεις, ε, οι εργαζόμενοι, δεν κερδίζουμε τίποτα με αυτές τις συμφωνίες. Το αντίθετο, χάνουμε πολλά από τα δικαιώματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, από ό,τι φαίνεται οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε θέλουν να μείνουν ανοιχτέ αυτέ τι αναφορέ, οπότε θα συνεχιστεί η συζήτηση. Δεν θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε ακόμη. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο για τρία λεπτά στου αναφέροντε και κατόπιν θα συνεχίσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά που ακούσαμε είναι σωστά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω και το λέω αυτό από βαθιά πεποίθηση και είμαι καλός Ευρωπαίος. Όσον αφορά το ISDS, τις προσφυγές των επενδυτών και την ε, νομοθετική συνεργασία, αυτά είναι πολύ επικίνδυνη πτυχή στις διαπραγματεύσεις και εάν περάσει τέτοιου είδους δημοκρατία, αυτό θα οδηγήσει σε τεράστιες αντιδράσεις. Και θα οδηγήσουν και σε πάρα πολύ ψηλό κόστος αν χρειαστεί να πληρώσουμε ε, αυτούς που υποβάλλουν προσφυγές, τους επενδυτές δηλαδή. Θα αφήσουμε ανοιχτή, ανοιχτές τις αναφορές αυτές και θα παρακολουθήσουμε την συνέχεια τέθηκε και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Δύο λεπτά μόνο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Δύο ήταν ερωτήσει που υπευλήθησαν πρώτα-πρώτα όσον αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών και ακριβώ όπως είπε ο αξιότιμο βουλευτής, εμείς δεχθήκαμε την ε, δικαστική απόφαση και λάβαμε τις αντίστοιχε δέουσες ε, αποφάσει για να συμμορφωθούμε, οπότε έχουμε τώρα ε, αυτήν την ε, πρωτοκόλληση στις 4 Εβδόμου της πρωτοβουλίας και ε, ε, ολοκληρώθηκε, μάλλον ξεκίνησε η επίσημη διαδικασία και η πρώτη διαδικασία που κρατά ένα χρόνο ξεκίνησε 10 Ιουλίου. Βεβαίω και μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και δεν πιστώθηκε αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αποτυπώνεται αυτό και στη, στο ψήφισμα αλλά επίσης και στην δικαστική απόφαση. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έλαβε όλα αυτά ε, όσον αφορά το τι συνέχεια τις αναφορές και ίσως έχετε υπόψη το ότι φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης για μεταρρυθμίσεις. Οπότε όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά έχουμε να σας πούμε προς το παρόν. Τώρα όσον αφορά τη διαδικασία επίλυσης των διαφόρων για να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο, ο κόσμος όσον αφορά ε, αυτό το, το δικαιοδοτικό όργανο για τις επενδύσεις λάβαμε υπόψη το βελγικό ψήφισμα αναλύσαμε το περιεχόμενο αλλά ακόμα δεν μπορούμε να δηλώσουμε τίποτα με μεγάλη προσοχή να εξεταστεί και μελετηθεί όλα αυτά θα υπάρξει σχετική απόφαση και όσον αφορά την ε, ΣΥΤΑ ξέρετε ότι υπάρχει προσωρινή ε, ισχύς και οριστικά θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία μόνο όταν όλα τα κράτη-μέλη με τα κοινοβουλία τους έχουν κυρώσει αυτήν την συμφωνία. Έχουμε το, τα κεφάλαια ε, για τις επενδύσεις και για το σχετικό δικαιοδικό όργανο τα οποία δεν τίθενται σε ισχύ, δεν ισχύουν και πρόκειται να συζητηθούν περαιτέρω. Και εν προκειμένου έχουμε διαφορετικές ε, αποφάσεις αλλά θεωρούμε ότι στο παρελθόν ε, είναι σύνομο σύμφωνα με αποφάσεις του, δικαστηρίου να υπάρξει ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τέτοιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αυτά σύμφωνα με την ε, νομολογία του δικαστηρίου, εφόσον όλα αυτά συνάδουν προς τις διεθνείς συμφωνίες. Αυτά, τυρμές αυτονομίας του κοινοτικού δικαίου και της ε, αρμοδιότητας της αποκλειστικής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα συνεχιστεί αυτή η πορεία, θα κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες του θέματος και φυσικά λαμβάνουμε υπόψη όλες τις ε, απόψεις αυτά. Πρόεδρε, ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, αγαπητοί συναδελφοί, το θέμα είναι περίπλοκο. Ο διάλογος συζήτηση θα συνεχιστεί και θα μείνουν ανοιχτέ οι αναφορές, αν συμφωνείτε. Κυρία Εύη. Κύριε, κάποιε πολιτικέ ομάδε έχουν ζητήσει να διαβιβαστούν στα κράτη-μέλη αυτές οι αναφορέ, τόσο ώστε να γνωστοποιηθεί το ότι έχει ξεκινήσει εδώ πέρα η ζήμαση και ότι όλα αυτά γίνονται με διαφάνεια στην Επιτροπή Αναφορών. Διαβίβαση από την Επιτροπή Αναφορών. Βάλε Περισσότερε πολιτικέ ομάδε θέλουν να γίνει, να εισταλεί αυτή η αποστολή. Ίσως όμως να περιλάβουμε και την επίσημη θέση της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου που ενέκρινε, συμφώνησε με την ΣΥΤΑ. Να μην στείλουμε μόνο αυτές τις αναφορές στα κράτη-μέλη να στείλουμε και την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου. Κύριε Μαριά. Ε, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ σημαντικό να αποσταλεί η επιστολή ενημέρωση στα κράτη-μέλη, διότι έχουμε μια διαδικασία ανοιχτή ως προς την επικύρωση. Και αν προσέξατε τι είπε η Κομισιόν, είπε ότι για να τεθεί σε οριστική εφαρμογή πρέπει να κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή τι θα γίνει πρακτικά. Αν δύο κράτη-μέλη το αμφισβητήσουν, η εφαρμογή προσωρινή από τώρα μέχρι τα επόμενα δύο χρόνια είναι παράνομη. Γι' αυτό λέω ότι έχει δημιουργηθεί μια παράνομα de facto κατάσταση. Άρα λοιπόν να πάει η επιστολή στα κράτη-μέλη και προφανώς δεν έχουμε αντίρρηση να εξηγηθεί και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία κατά την άποψή μας είναι εξίσου παράνομη. Διότι το να εφαρμόσεις προσωρινά μια συμφωνία που πιθανόν να ακυρωθεί όταν θα έχουν δημιουργηθεί δυσμενή αποτελέσματα, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει εφαρμογή σοβαρή του κοινοτικού δικαίου. Αλλά α αποσταλεί και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι την είχαμε καταψηφίσει. Rendben, tehát, rendben, tehát Ωραία. Θα ενημερώσουμε τους εκπροσώπους των κρατών μελών με επιστολή. Θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τη θέση και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου μέχρι στιγμής. Θα τους ενημερώσουμε ότι έχουν προκύψει αμφιβολίες σχετικά με την συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Το κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια μάλλον δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν αυτή τη συζήτηση τόσο ή άλλως. Δεν θέλω να ε, δώσω περισσότερη συνέχεια στο θέμα, αλλά επειδή πολλέ από τι αναφορέ είχαν να κάνουν με τη διαφάνεια, προτείνω να σταλεί επιστολή στο Συμβούλιο ζητώντα του ε, να ε, δημοσιεύσουν τι διαπραγματευτικέ εντολέ κλπ. Διότι αυτό φαίνεται να είναι βασικό μέτρο για να βελτιώσουμε την διαφάνεια στην εμπορική πολιτική. Ε, ωραία, θα στείλουμε τις επιστολές αυτές. Αν συμφωνείτε όλοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη αναφορά. 1804 κάθετος 2013 σχετικά με την ένδειξη Made in EU. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ντομάτζη από την, τον κύριο Λεβάτζη Μάλλον βρίσκεται εδώ αναφέρον ο κύριος... Ο κύριος Παύλο Λάβατσι... από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ένδειξης Made in EU σχετίζεται με την ε, πρόταση 2013 κάθετος 78 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. κατάφαστα θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στα τρόφιμα και στα μη εδόδημα προϊόντα. Για τα μη εδόδημα προϊόντα η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτεί αυτή τη στιγμή η χώρα προέλευσης να αναγράφεται στο προϊόν. Ωστόσο, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αναφέρουν την προέλευση του προϊόντος και ο θελός. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Για παράδειγμα, ότι οι πληροφορίες πρέπει να είναι αληθείς. Ε, σύμφωνα με την ε, οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Υπάρχει όμως η δυνατότητα για οικονομικό φορέα να αναφέρει για τα μη εδόδημα προϊόντα είτε το ένα είτε το άλλο. Δηλαδή είτε την ένδειξη Made in EU ή ε, τη χώρα στην οποία κατασκευάστηκε το, το κράτος μέλος. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέο κανονισμό ε, προβλέπει για να ενισχυθεί η ταυτοποίηση και η χνηγασιμότητα των προϊόντων ε, να είναι υποχρεωτική η ένδειξη της χώρας καταγωγής. Ωστόσο, ο οικονομικός φορέας μπορεί να αναφέρει είτε το κράτος μέλος, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τα τρόφιμα, η βασική αρχή είναι ότι η καταγωγή παραμένει προαιρετική, εκτός εάν η παράληψή της ε, μπορεί να παραπλανήσει τον ε, καταναλωτή. Οι διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων ε, περιορίζονται σε κάποια προϊόντα, όπως είναι το κρέας που έχει τυχή επεξεργασίας, το μεταποιημένο κρέας. Όσον αφορά την επεξεργασία σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Εκτός από το μέλι ε, και το μη επεξεργασμένο κρέας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η σήμανση Made in EU επιτρέπει Ε, την ε, αναφορά όλης της αλυσίδας παραγωγής ε, που είναι χρήσιμη πληροφορία για ένα προϊόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γιάροσλαβ. Βαλέσα. Μ' αρέσει το σήμα με την γιου. The product uh, is kept with uh, certain standards. αυτό σημαίνει ότι το προϊόν διέπεται από κάποια πρότυπα, κάποια επίπεδα. Το χρειαζόμαστε αυτά τα στάνταρ, το περιβάλλον, κοινωνικά, για διάφορα προϊόντα. Οπότε, όταν βλέπω αυτό το σήμα, τότε αυτό με κάνει να αγοράσω το προϊόν. Για διάφορα προϊόντα. Επομένω, θεωρώ ότι πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά, γιατί νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να υπάρχει αυτή η επισήμανση. Κύριε Μαρία. Νομίζω ότι από την τοποθέτηση της Κομισιόν αναδεικνύονται ορισμένα σοβαρά ζητήματα. Πριν από την προηγούμενη Πέμπτη ήμουν στην Επιτροπή Γεωργίας και εκεί συζητούσαμε για το μέλι. Ήρθε λοιπόν ένα συνάδελφος από τη Βουλγαρία και κατήγγειλε πολύ σωστά ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πρόσμιξη μελιού το οποίο εισάγεται από την Κίνα με βουλγαρικό μέλι και στο τέλος λέει μέλι Βουλγαρίας και μετά αυτό είναι made in EU. Αυτό το μέλι επίσης σύμφωνα με καταγγελίες που έχουμε από Έλληνες παραγωγούς το βουλγαρικό έρχεται στην Ελλάδα και γίνεται και αυτό ανάμιξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι απαιτείται η σήμανση, απαιτείται η εχνηλασιμότητα και ακόμη και στο μέλι ή στο κρέας που είπε η Κομισιόν που υπάρχει υποχρέωση και πάλι βλέπουμε να γίνεται κομπίνα, να γίνεται απάτη, να έχουμε προϊόντα μαϊμού. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα για να γνωρίζουμε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας των τροφίμων. Αν πράγματι είναι ευρωπαϊκά ή έχει γίνει ήμι επεξεργασία σε τρίτες χώρες και μετά εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουν και μια σφραγίδα ευρωπαϊκή. Για δε τα βιομηχανικά προϊόντα, τα περισσότερα πλέον ήμι παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε τρίτες χώρες και απλά έρχονται την τελευταία στιγμή στο τελευταίο στάδιο και γίνεται μια μικρή επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνει φραγίδα EU. Άρα λοιπόν πρέπει να τα προσέξουμε όταν λέμε EU να εννοούμε EU Δηλαδή να εννοούμε ότι πράγματι έχει γίνει η διαδικασία παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά πρέπει να υπάρχει η πλήρης διαδικασία της σήμανσης, της ίχνη λασιμότητας για να μην δημιουργούνται προβλήματα ως προς τους καταναλωτές. Διότι πρέπει να προστατεύονται, υπάρχουν θέματα υγείας, υπάρχουν θέματα απάτης κλπ. Επομένως νομίζω ότι αυτή η αναφορά είναι σημαντική, μας έδωσε ευκαιρίες και ίσως ε, είναι μια ευκαιρία εδώ στην Επιτροπή μας να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε, όπως λέει ο συνάδελφος ο Γιάννουσλαφ την αναφορά, αλλά να τη στείλουμε για ενημέρωση και σε αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου μας. Δηλαδή είτε στην Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων, είτε στην Επιτροπή για θέματα βιομηχανίας, για να πάρουν ένα feedback και να έχουν έτσι και αυτή καλύτερη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Αφού δεν θέλει άλλο το λόγο, τότε σας προτείνω το εξή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που άκουσαμε τον κύριο Μαριά. Αυτό αφορά όμως την προστασία του καταναλωτή. Για να αναφέρει η ένδειξη ελληνικό μέλι, αλλά περιέχει άλλο μέλι μέσα, αυτό αποτελεί μια απάτη. Ακόμα και λέει Made Τέλος πάντων, ε, ας κλείσουμε την αναφορά, αλλά στείλουμε στην ΙΜΚΟ όλα τα σχετικά στοιχεία. Συμφωνείτε? Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, η επόμενη αναφορά είναι η παριθμόν 0709 κάθος του 2016. Αφορά ένα πρόβλημα μεταξύ τελικών τραπεζών και τη Εθνική Εποπτική Αρχή. Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριο Γκαϊτάνο Βίλνο βρίσκεται εδώ και του δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι θα πρέπει να μην ξεχνάμε τον ε, Πυθαγόρα όσον αφορά τη βελτίωση της Ζωή της ποιότητας ζωής του κόσμου και θα θυμάστε τι θυσίε έχουν γίνει για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Γιατί εδώ ήρθα και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο μια που πρέπει να σας πω ότι απευθύνομαι στην ε, λογική σας όσον αφορά τους νόμους, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ακριβώς την ευημερία του κόσμου. Αλλιώς κάτι πάει στραβά. Στην ε, Ιταλία από το 2015 μέχρι σήμερα έχουμε από πλευράς του κράτους 70 δις ευρώ που έχουν παρασχεθεί στις τράπεζες με πάρα πολλές ε, φάνταστες δικαιολογίες. Έχει υιοθετηθεί μια εποπτική πολιτική και έχουν ξεχάσει οι υπεύθυνοι τα συμφέροντα των αποταμιευτών. Έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Οι Ιταλικές τράπεζες έχουν ε, ε πωλήσει τοξικά προϊόντα και έτσι έχουν καταστραφεί πάρα πολλά φυσικά πρόσωπα αλλά και οι μικρές εταιρείες από την τράπεζα Βένετο και άλλη μία και είναι λογικό να λάβουμε υπόψη αυτά τα 300 τόσα εκατομμύρια τα οποία είναι οι αποταμιεύσεις μας και είναι αποταμιεύσεις μια ζωής τι είναι αυτό το οποίο έγινε ποιος φταίει φταίμε όλοι από λίγο και είμαστε και μέλος, μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης οπότε εγώ τώρα τι κάνω. Πρέπει τώρα να ελέγχω τις τράπεζες, την ομιμότητα των ενεργειών τους και την ποιότητα των προϊόντων τους. Οπότε τελικά θα πρέπει με τα λίγα που ξέρουμε και κυρίως με το ανθρώπινο συνέστημα να σταθμίσουν τα πράγματα, να δούμε ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Η κυβέρνηση Αμάτο από το 1992 ε, μετέφερε στην ε, Τράπεζα της Ιταλίας την εποπτεία των ε, τραπεζών. Και σήμερα έχουμε αυτή την τράπεζα που είναι ανώνυμη εταιρεία. Αυτό γίνεται κατά παράβαση του ίδιου του καταστατικού της τράπεζας της Ιταλίας. Θεωρώ ότι αυτό αρχεί, ότι δηλαδή το εποπτικό όργανο είναι η διοκτησία των ίδιων των τραπεζών που ελέγχει. Αυτό δεν είναι εγγύηση αμεροληψίας. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2005 στο Λέτσε έκρινε ένα δικαστήριο στο Λέτσε ότι έχει ε, βλάψει κάποιον ε, αποταμιευτή και τον αποζημίωσε. Και έχουμε αυτήν την ε, απόφαση που αφορά την περίοδο μέχρι το 2003 και έχει θεωρηθεί ότι συνολικά έχει παραβλάψει η τράπεζα τους πολίτες κατά 5 δισεκατομμύρια συνολικά. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία που όμως έχει μονοπωλιακό ρόλο δεν υφίσταται κρατικό έλεγχο. Και έχει και την ε, αρμοδιότητα του ελέγχου όλων των τραπεζών, των ιδιωτικών. Θα μπορούσαμε επί ώρες να μιλούμε για τους νόμους και για το πώς θα μπορούσε κάτι που είναι αδιανόητο να έχει την ε, εικόνα της νομιμότητας. Οπότε και τώρα σε εσά απόκειται αυτό το οποίο ζητούμε. Κατά τη γνώμη σας, είναι λογικό το εποπτικό όργανο να είναι μια ανώνυμη εταιρεία και αυτές οι μετοχές αυτής της ανώνυμης εταιρείας να ανοίγουν σε ίδιες στις τράπεζες. Πρόκειται για ληστείες βάρος της Ιταλίας, για ληστείες βάρος της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Τσέζαρη, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, αυτό που έχουμε να πούμε γίνονται γύρω από δύο άξονες. Πρώτα-πρώτα σκεφτόμαστε αντίστοιχα το πώ είναι δομημένη αυτή η αναφορά που πρώτα-πρώτα, ε, όπως την ακούσαμε στην προφορική ανάπτυξη, που αφορά την διακυβέρνηση της Τράπεζας Ελλάδα και από την άλλη μεριά τον ρόλο του Κόντσομπ, τις πληροφορίες δηλαδή που αφορούν τα δελτία, τα, τα, τα προσπέκτους για τους επενδυτές. Όσον αφορά τώρα την διοίκηση διακυβέρνηση της τράπεζας, θεωρούμε ότι οι κοινοτικέ διατάξεις που αφορούν αυτό το ζήτημα και ιδίω το άρθρο 4 της οδηγίας 37 του 13 ορίζουν ότι είναι υποχρέωση του κράτους να παράσχει εγγυήσεις ότι δηλαδή το εποπτικό όργανο έχει την ανεξαρτησία και οικονομική ανεξαρτησία από τους ελεγχομένους. Η Τράπεζα της Ιταλίας ιστορικά είχε δομή ανώνυμης εταιρεία. Δεν είναι η μόνη ε, τράπεζα που είναι ανώνυμη εταιρεία και η μόνη που έχει βουτικές αρμοδιότητες στην Ευρώπη όντας ανώνυμη εταιρεία και αυτού του είδους η μορφή η εταιρική δεν θεωρήθηκε ότι έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της ανεξαρτησίας και με την λειτουργία της τράπεζας ως εποπτικής αρχής και αυτά κατοχυρώνονται στην Ιταλική νομοθεσία και βεβαίως και υπήρξε και νομοθεσία που διέπειτα τις τραπέζες και έχουμε το νομοθέτημα ε, υπαριθμών 5 του 2014. Εκεί ρητά προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν μπορεί να αναμειχθεί στις εποπτικές λειτουργίες της τράπεζας. Επομένως, επαναλαμβάνω, λάμβοντας και υπόψη άλλα μοντέλα εποπτείας στην Ευρώπη. Δεν θεωρήθηκε ότι υπάρχει εδώ ε, σύγκρουση ε, με την αρχή της εξαρτίας της τράπεζας. Αυτό βεβαίω αυτό δεν αποκλεί να υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις, υπάρχουν συγκεκριμένες ποινικέ ευθύνες. Ακριβώς όπως την περίπτωση που μας ανέφερε ο αναφέρον. Ε, δεν μπορούμε όμως ε, σε αυτό να παρέμβουμε γιατί αυτό είναι θέμα εθνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό και περιορίζομαι στα της διακυβέρνησης, διοίκησης της τράπεζας. Και επαναλαμβάνω ότι η εταιρική μορφή της τράπεζας δεν διαφέρει από τις άλλες ε, εποπτικές ας πούμε τράπεζες της Ευρώπης. Και έχοντας και το νομοθέτημα του 2014 δεν θεωρείται ότι υπάρχει σύγκρουση ε, με την αρχή της ανεξαρτησίας Επίσης είχαμε αναθεώρηση του καταστατικού της τράπεζας κατόπιν της νομοθεσίας. Η ΔΕ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει αποφανθεί θετικά για το καταστατικό της τράπεζάς μας και για την ανεξαρτησία αυτής και για τον ρόλο της ως εποπτικής αρχής. Και δίνω τη σκητάλη στον συνάδελφο. Καλημέρα σας. Ρώση και Φιωρέλο ονομαζόμαστε. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο άξονα της παρέμβασης, όσον αφορά δηλαδή το αίτημα προς τις ευρωπαϊκές αρχές για να ερευνήσουν και να επιβάλλουν κυρώσεις ε, όσον αφορά τις ευθύνες της Κόντσομπ. Έχουμε δεδομένη την οδηγία 71 του 2003 για το προσπέκτους και αναφερθήκατε ε, σε κάποια ανακοίνωση της Κόνσοπ του 2009, ένα ενημερωτικό σημείωμα επίσης του 2011, σε αυτά αναφέρθηκε η αναφορά. Η ανακοίνωση του 9 της Κόνσοπ αναφέρει το ότι χρειάζεται να υπάρχουν τα σενάρια επικινδυνότητος κάποιων προϊόντων. Αυτό υπέρ του πελάτη. Να ξέρει επομένως τι κινδύνους διατρέχει. Και έτσι η Κόντσομ δεν θέσπισε δεσμευτικό κανόνα για αυτά τα σενάρια επικινδυνότητας στα δελτία, στα προσπέκτους με την εσωτερική με το ιστορικό σημείο του 2011 η Κόνσοπ ε, εμένει και αυτό λέει και η αναφορά σε σχέση με τα σενάρια επικινδυνότητας. Πολλοί από τα μία αυτές εζημιώθηκαν διότι τοποθέτησαν τα χρήματά τους σε κάποια προϊόντα τραπεζικών ιδρυμάτων που αντιμετώπισαν δυσκολίες. Και το θέμα είναι κατά πόσον υπήρχε ή όχι επισήμες των κινδύνων στο προσπέκτους η, Επιτροπά, η Επιτροπή συγγνώμη, ως φύλακας των συνθήκων παρεμβαίνει όποτε τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν ορθώς το κοινοτικό δίκαιο ή όταν υπάρχει σύγκρουση εθνικής με κοινοτική νομοθεσία. Οπότε αυτή η ανακοίνωση του 2009 της Κόνσοπ δεν αντιβαίνει στις αρχές της ε, οδηγίας 71 του 2003 για τα προσπέκτους ούτε στον κανονισμό 809 του 4. Οπότε αυτά τα οποία αναφέρονται εις βάρος της Κόνσοπ δεν είναι αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής και αφορούν ε, την ορθότητα της εφαρμογής της σχετικής οδηγίας στην Ιταλία. Ο Πρόεδρος. Είναι ένα θέμα αρμοδιότητα και νομίζω ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Θέλετε το λόγο κύριε Βάλη, εντάξει, για δύο λεπτά. Πολύ γρήγορα πρέπει να σα τα πω αφού δύο λεπτά. Ευχαριστώ τον αναφερθώ δεν τον γνωρίζω, αλλά συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα μα είπε. Το θέμα είναι ακριβώς ποιοι είναι οι κάτοχοι των μετοχών της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Ε, ε, Πρόκειται για την συμμετοχή των ιδιωτών, ε, αλλά είπαμε ότι πάνω το 50% ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει άλλη τέτοια τράπεζα στην Ιταλία, πάνω από 50% είναι αυτή. πρόκειται για σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άπαξ και ο ελεγχόμενος, ο εποπτευόμενος συμμετέχει σε με τέτοιο ποσοστό ε, επί της Τράπεζας Ιταλίας που είναι η εποπτική αρχή. Τώρα, όσον αφορά την Κόνσοπ και αυτή την σύγκρουση συμφερόντων, ε, ακούσαμε τι γίνεται, ακούσαμε ε, τι ενδείξεις υπάρχουν και πώς υπάρχει παραπίση της αλήθειας, πώς οι επενδυτές δεν ειδοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Υπέστησαν εξαπάτηση. Και δεν είναι θέμα συγκεκριμένων μεμονωμένων περιπτώσεων. Ήταν κάτι που έλαβε χώρα ευρέως και ευνηδιαστικά. Και λέει εδώ πέρα ότι δεν είναι θέμα σύγκρουση συμφερόντων και συμμετοχή μόνο των ιδιωτικών τραπεζών στην Τράπεζα τη Ιταλία. Πρόκειται για μια κατάσταση στην Ιταλία οπότε δεν, δεν τηρήθησαν, δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα των καταναλωτών οι οποίοι εξυπατήθησαν. Θα πρέπει η Κεντρική Τράπεζα ακριβώς λόγω της λειτουργίας της θα πρέπει να είναι κρατική η Κεντρική Τράπεζα. Και εδώ έχουμε σύγκρουση συμφέροντων. Και ακριβώς το λέει η σχετική οδηγία. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι είναι ανεξάρτητες οι ελεκτικές εποπτικές αρχές και να υπάρχουν όλες οι εγγύες ανεξαρτησίας για να εκτελούν το καθήκον αρμοδιότητά τους. Αυτό ισχύει και για την Ιταλία και στον υπόλοιπο κόσμο. Μα δώστε μου παραδείγματα εταιριών κάπου στον κόσμο, κεντρικών κρατικών τραπεζών, όπου ε, το πίνεσφο του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε ιδιώτες. διότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας αποδεικνύεται ότι έχει μετόχους άλλες τράπεζες και ιδιώτες. Το ίδιο ισχύει και για την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει νομίζω και για την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κεντρικές τράπεζες οι οποίες στην πλειοψηφία του μετοχολογίου τους ανήκουν σε ιδιώτες. Στην Ελλάδα μάλιστα το κράτος δεν επιτρέπεται να έχει πάνω από 5% συμμετοχές. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Διότι οι κεντρικές τράπεζες παίζουν σοβαρό ρόλο πλέον στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης. Στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν ομόλογα ιδιωτών είτε εταιριών είτε τραπεζών και επομένως υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Και επειδή έχουμε ρωτήσει επανειλημμένα τον κύριο Ντράγκη λεπτομέρειες για το ποιες μετοχές αγοράζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του QE και μας έχει απαντήσει ότι δεν μας δίνει λεπτομέρειες για το τι αγορές έχουν κάνει οι κεντρικές τράπεζες είτε η Τράπεζα της Ελλάδος που είχα ρωτήσει εγώ που διέθεσε 17 δισεκατομμύρια ευρώ η Τράπεζα της Ελλάδος και αγόρασε ομόλογα στην ποσοτική χαλάρωση. Την ίδια ερώτηση είχε κάνει και ο κύριος Βάλλη για την Ιταλία. Την ίδια ερώτηση είχαν κάνει και συνάδελφοι Ισπανοί. Επομένως εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Και πρέπει να το δούμε. Και η πρότασή μου είναι ότι πρέπει η αναφορά να έρθει στην οίκον για να κάνουμε μια συζήτηση σοβαρή, διότι άλλη ήταν η εποχή όταν πρωτοξεκίνησε το ευρωσύστημα και υποτίθεται ότι έγινε δεκτό από την ECB ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος και η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας και του Βελγίου μπορούν να είναι στο χρηματιστήριο. Ήταν μια άλλη εποχή. Τώρα με το ρόλο που παίζουν στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης πρέπει να δούμε την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων και επομένως το θέμα να παραμείνει ανοιχτό Δεύτερον, να έρθει για ενημέρωση στην Επιτροπή Οικονομικών της, ε, του Ευρωκοινοβουλίου και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Γιατί υπάρχουν θέματα σύγκρουση συμφερόντων σίγουρα και πρέπει να τα δούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να έχουμε διδαχθεί από την τελευταία οικονομική κρίση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ε, πολλά για την τραπεζική εποπτεία και γι' αυτό και έχουμε εγκρίνει τόσο πολλούς νόμους, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξαναέχουμε μια τραπεζική κρίση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προκείμενο, λέει ότι δεν παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Κομισιόν ε, και αν εδώ δεν πάει κάτι καλά, αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Και εγώ θα ήθελα να, να πω ότι πραγματικά ε, και εγώ ε, σίγουρα έχω ε, ως ε, μέλος της Επιτροπής Αναφορών πολύ δουλειά και δεν έχω εμβριθώς μελετήσει. Γι' αυτό εμπιστεύομαι τον κύριο Μαριά και πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την άποψή του. Και σίγουρα υπάρχει το οικονομικό ζήτημα εδώ, είναι τα χρήματα Πιστεύω ότι καλά κάναμε μεν και φροντίσαμε τις τράπεζες να τις γλιτώσουμε από την κρίση και να τις διασώσουμε, αλλά τώρα πρέπει να δούμε στην προκειμένη περίπτωση τι γίνεται. Συμφωνώ με τον κύριο Μαριά. Θα ήταν ίσως καλό να το αναλάβει μια επιτροπή η οποία έχει αρμοδιότητα επί των θεμάτων αυτών, ε, αλλά συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Μαριάς. να μην γίνει πάλι κάτι που θα οδηγήσει σε μια κρίση που κανένας δεν θα ήθελε στην Ευρώπη. Ακούστε, η κατάσταση έχει ως εξή. Ίσως να δεχτεί και ο κύριος Μαριάς αυτό που θα πω. Πρόβλημα υπάρχει, εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το θέμα. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ έχει αρμοδιότητα όμως και είχε στις 19 Ιουλίου μια μακροσκελέστη συζήτηση επί του θέματος. Αποφάσισε ότι στην Ιταλία εναπόκειται να λύσει το ζήτημα. Είναι εθνικό θέμα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και σας συστήνω να κλείσουμε την αναφορά, όμως να την ε, στείλουμε ενημερωτικά την υπόθεση αυτή και στην ε, Κεντρική Τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να την προειδοποιήσουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν αυτό μπορείτε να το αποδεχθείτε. Κοιτάξτε, η Ευγεία το λέει ότι πρόκειται αυτό να ρυθμιστεί κατά αυτόν τον τρόπο, ακριβώ όπω μα είπε η Επιτροπή απαντώντα στον αναφέροντα και λέει ότι πρέπει τα κρατημέρια να εξασφαλίσουν το ότι οι αρμόδιε ε, προ εποπτεία αρχέ θα έχουν την αναγκαία ανεξαρτησία, ούτω ώστε να ασκήσουν αρμοδιότητέ του. Ε, ναι, ε, το καταλαβαίνω, αλλά άπαξ και έχουμε κάποια εταιρεία όπου κατά το 100% ε, υπάρχει τέτοια ε, συμμετοχή των ιδιωτών, μα τότε πώς θα μπορέσει να κάνει την εποπτεία. Να, η σύγκρουση των συμφέροντων. Επομένω, θα πρέπει τώρα που έχουμε αυτή την αναφορά κάτι να κάνουμε, αλλιώς ενεργούμε παράλογα. Πρόεδρος. Ακούστε. Η αρμόδια επιτροπή, η ΕΚΟΝ, που ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε αρμοδιότητα εμείς για κάποια περαιτέρω ενέργεια. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα να κλείσει η αναφορά, να σταλεί προειδοποίηση στην ΕΚΤ και να πω στους αναφέροντες ότι αν υπάρξει κάτι νέο μπορούν να επανακαταθέσουν μια νέα αναφορά για το θέμα αυτό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, αλλά προς το παρόν κάτι άλλο με την παρούσα αναφορά δεν μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο, που είναι η έκθεση για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος του συγκεκριμένου. Δηλαδή ποιο είναι το ερώτημα σήμερα. Το ερώτημα είναι το εξής. Είναι δυνατόν να υπάρχουν εθνικές κεντρικές τράπεζες όπως είναι στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στο Βέλγιο που οι μετοχές τους να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και να έχουμε ιδιώτες μετόχους. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και σε αυτό εμείς θέλουμε να γίνει συζήτηση σοβαρή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το μοντέλο του ευρωσυστήματος. Επομένως θεωρώ ότι μετά τη συζήτηση που κάνουμε πράγματι να στείλουμε την αναφορά στην ECB αλλά να την ξαναστείλουμε στην ECON με το ερώτημα αυτό ότι πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει το ευρωσύστημα σωστά όταν ορισμένες εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια άλλη συζήτηση διαφορετική την οποία πρέπει να κάνουμε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και εγώ και ο κύριος Βάλλη που είμαστε μέλη να το θέσουμε αυτό το θέμα. Αλλά να υπάρχει η αναφορά να έχει σταλεί και να υπάρχει το ερέθισμα για συζήτηση. Και, και, Αγαπητέ συνάδελφε, η αναφορά στις 19 Ιουλίου κοινοποιήθηκε στην ε, Οικονομική Επιτροπή. Όμως, είπαμε ότι δεν έχει την ε, κυρίως αρμοδιότητα Πάντως μπορεί να υποβάλει νέα αναφορά ο θυγόμενος. Κυρία Μπεθέρα. Παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Ακούστε. Πράγματι, θα είμαι σύντομη γιατί έχει τελειώσει και ο χρόνος και θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς οι οποίοι είναι εδώ. Ελπίζω να μα δώσουν λίγο χρόνο παραπάνω. Για να συζητήσουμε κάτι που όλου μα ανησυχεί. Και νομίζω ότι είναι και μια από τι πιο σημαντικέ ε, κοινοβουλευτικέ πρωτοβουλίε. Ε, αυτό για την Επιτροπή Αναφορών Έκθεση για την Ιθαγένεια. Είναι μια έκθεση η οποία διεξάγεται ε, μία φορά στα τρία χρόνια. Ελπίζω η, τρία, ε, η τρίτη να είναι και καλή και να έχουμε την τελική έκθεση η οποία θα βάλει τις βάσεις, ε, θα βάλει τα θεμέλια. Όταν ιδίω εορτάζουν την 25η επέτειο από τη συμπερίληψη της Ιθαγένειας στην συνθήκη του Μαστρίχτ, τότε άρχισαν να γίνεται λόγος για Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα ήθελα εγώ να σας αναφέρω κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό το έγγραφο μπορείτε να βάλετε και τροπολογίες. Είναι πολύ σαφή ε, η θέλησή μας και υπάρχει συνένεση να εστιάσουμε στα κεντρικά σημεία. Στη Λίμπε υπάρχει συνεισηγητής ε, που βρίσκεται ακριβώς ε, στην ίδια γραμμή και με μένα. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι σε ό,τι αφορά τη σκοπιμότητα που θέλει να εξυπηρετήσει αυτή η έκθεση είναι να αντιμετωπίσει τι άνευ προηγουμένου προκλήσεις και δει τι επιπτώσεις ε, που θα έχει το Brexit για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Επίση, άλλο σκοπό είναι η ηθαγένεια ε, να έχει μια σαφή αξία για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι αναγνωρισμένα και έχουν μεγάλη αξία, Όπω είναι η ελευθερία κυκλοφορίας. Αλλά το 20% μόνο των πολιτών ασκεί αυτό το δικαίωμα. Όλοι οι Ευρώποι πρέπει να νιώθουν ότι επειδή ακριβώ έχουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια μπορούν να απολαμβάνουν αυτή και αυτό να αποτελεί κίνητρο. Ποια είναι τα βασικά μηνύματα τη έκθεση. Ποιο είναι ο ε, η σπονδυλική στήλη αν θέλετε, είναι η μη διακριτική μεταχείριση. Δηλαδή θέλουμε να πετήσουμε η οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων που είναι σε ένα σερτάρι 10 χρόνια λόγω των μελών του Συμβουλίου, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, να κινητοποιηθούμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μέσα στο σχέδιο Γιούνκερ και θα πρέπει η Κομισιόν να το ενεργοποιήσει. Ποιοι είναι οι πυλώνε στου οποίου εδράζεται η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είναι η ισότητα, δηλαδή καμία διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας, ε, ε, πεποίθησης, ε, γλώσσας. Το δικαίωμα υποβολής αναφορών υπάρχει αυτό το δικαίωμα ε, πάνω στο οποίο δράζεται και η Επιτροπή μας και η ίδια η έκθεση και η συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή, που σημαίνει ψηφίζει χωρίς εμπόδια, κυρίως ελεύθερα, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και άλλα θεσμικά όργανα, αλλά κυρίως το Κοινοβούλιο, στο πλευρό των πολιτών. Σε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να υπάρχουν και υπάρχουν γραφεία υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του Κοινοβουλίου τουλάχιστον. Και θα πρέπει αυτό να είναι ε, μια ενιαία θηρίδα, ένα one-stop shop για τους πολίτες. Όλα αυτά οδηγούν στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής, ενός ευρωπαϊκού χώρου ε, ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας. Σε ό,τι αφορά τις ε, προθεσμίες. Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Υπάρχουν τρεις γνωμοδοτήσεις από τις επιτροπές ΑΦΚΟ, ΚΟΥΛΤ, ΦΕΜ και η προθεσμία για την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας είναι 22 Νοεμβρίου. Επικοδομητική είναι η διάθεσή μας και πραγματικά στην Επιτροπή Αναφορών θέλουμε να δώσουμε ένα σαφή χαρακτήρα, σαφές πλαίσιο για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους που θα με συνοδεύσουν σε αυτό το μονοπάτι ότι θα κάνουν και αυτοί πάντο δυνατόν. Εγώ θέλω εδώ να πω ότι αυτός ο στόχος, δηλαδή ότι θέλουμε να γκρίνουμε ένα κείμενο στέρεο, που θέλουμε να εγκριθεί και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο, αυτό είναι ο στόχο και πιστεύω ότι μπορούμε να τον πετύχουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνεί. Είμαι σκιώδης εισηγήτης στην Επιτροπή Αναφορών. Ο συνάδελφός μου κ. Σόγκοτη είναι στη Λίπε και το ΕΛΚ στηρίζει το έγγραφο αυτό. Νομίζω ότι όλοι το στηρίζουν. Νομίζω ότι κάθε ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα να διαμορφώσει θέση. Και τρεις η ώρα στις 28 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στις 22 Νοεμβρίου εδώ στην Επιτροπή Πέτη. Otherwise, I make a proposal because we... Έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, Αλλιώ προτείνω, επειδή είμαστε ευέλικτοι, να ξεκινήσουμε στι 3 με το θέμα αυτό, ώστε να δώσετε το λόγο στους σκιώδεις για να πούνε λίγα λόγια για την έκθεση αυτή, διότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Καταλαβαίνω ότι οι διερμηνείς πρέπει να φύγουν. Θα ξεκινήσουμε στις 3 η ώρα. Δέκα λεπτά να μας δώσετε στην αρχή της συνεδρίασης για να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω στην έκθεση αυτή. Θα ενημερώσω την κυρία Βίκστρομ για το θέμα αυτό. Από εκείνη εξαρτάται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. The situation is very critical. <laughs> Thank you.